εγκρίθηκαν 10 έγγραφα, 10 πράξει σύμφωνα με την κανονική ε, νομοθετική διαδικασία, οι οποίε και θα δημοσιευθούν στα πρακτικά τη συνεδρία και για ένα διαδικαστικό από τον κύριο Στούγκαρ. Έχουμε. Ja, voorzitter, dank u wel. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Αυτό που πραγματικά με συγκίνησε στην ομιλία σα είναι το γεγονό ότι βάζετε στο επίκεντρο τη δημοκρατία. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι κατανόητο πραγματικά το γεγονό ότι στη διάσκεψη των Προεδρών αποφασίστηκε να μην γίνει συζήτηση για το Ολλανδικό δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στι 6 Απριλίου. Το γεγονό ότι αγνοείται το δημοψήφισμα και το αποτέλεσμά του αποτελεί μια σφαλιάρα ε, κατάμουτρα στους ε, Ολλανδούς. Είναι μια ε, ευκαιρία που χάνουμε να δείξουμε σεβασμό στους Ολλανδούς. Είναι μια ευκαιρία που χάνουμε για το μέλλον, γιατί όλο και πιο συχνά θα έχουμε τέτοια δημοψηφίσματα και εξ όσων κατάλαβα πολλά προετοιμάζονται και για το TTIP. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στούγα. Η δημοκρατία σημαίνει ότι γίνονται και πλειοψηφικέ ε, ψηφοφορίες και η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίστηκε πλειοψηφικά να μην ακολουθήσουμε το αίτημα της ομάδας σας. Δημοκρατικά. Λοιπόν, ε, ο Πρόεδρος ε, και τα υπόλοιπα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων απερίψαν την πρότασή σας. Αυτή είναι πραγματικά ένα, αυτό είναι ένα βίωμα, κάτι που ζούμε ω δημοκράτε. και σήμερα προσπαθήσατε να το ξαναβάλετε στην ημερήσια διάταξη, αλλά τέτοια αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται εντό συγκεκριμένων προθεσμίων και δεν το πράξατε αυτό. Το υποβάλλατε μετά την λήξη τη προθεσμία. Δεν τηρήθηκε η προθεσμία. Και τώρα περνάμε. Ο Πρόεδρε, εχθές ε, είχαμε τις ε, ανοιχτές ε, πύλες και ήταν πολύ ευχάριστο. Έγινε μια πραγματική συζήτηση, εξαιρετικά ευχάριστη. Διάφοροι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ήρθαν φορώντας μαντήλα. Αυτό πραγματικά με σόκαρε βαθύτατα. Θα ήθελα να αποφασίσετε όταν στο μέλλον θα γίνουν τέτοιε μέρες με ανοιχτών ε, πυλών εδώ στο Κοινοβούλιο να υπάρχει, να, είναι, να μην θεωρείται αυτονόητο ότι οι γυναίκες ε, που φορούν μαντήλα μπορούν να μπαίνουν σε αυτή την αίθουσα χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσετε στην επόμενη τέτοια ευκαιρία μαρτυρία που θέλουμε να κάνουμε για την κοσμικότητα και την ελευθερία δεν δέχονται τέτοιες συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και περνάμε τώρα στο σχέδιο εργασία. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού ε, αποφασίστηκε η ημερήσια διάταξη, λάβατε το σχέδιο ημερήσια διάταξη, δεν ξέρω για σήμερα, αν υπάρχουν αντιρρήσει. Δεν έχω λάβει αντιρρήσει σε κάθε περίπτωση ούτε για σήμερα, ούτε για την Τρίτη. Για την Τρίτη τώρα, κύριε Σασόλη. Ε, κύριε Πρόεδρε, λαμβάνουμε αυτές τις μέρες πάρα πολλά νέα όσον αφορά για την ε, γιορτή της Ευρώπης. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Ευρώπη όπου υπάρχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά για τους οποίους δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μέρες γιορτής. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φιλοξενούμενοι της Ευρώπης. Τα νέα μας τα οποία έχουμε από περιοχές όπως αυτή της Ιδωμένης είναι νέα τα οποία είναι πολύ ανησυχητικά. Μιλάμε όλο και περισσότερο για δυσκολίε που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα. Μιλάμε όλο και περισσότερο για συνθήκε υγιεινείς οι οποίες είναι πραγματικά παράδεκτες και αβάσταχτες. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουμε να τιμήσουμε ακριβώς τις αρχές που μας υπενθυμίσατε εσείς στην εισαγωγική σας παρέμβαση, που είναι αρχές πάρα πολύ σημαντικές, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επισκεφθεί τους καταβλισμούς των προσφύγων στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, Ήμασταν στην ημερήσια διάταξη. Αυτό συζητήσαμε. Συζητήσαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και για αύριο, για την Τρίτη. Δεν καταλαβαίνω εκ πρώτη όψεω τι έχει να κάνει η παρέμβασή σα με την ημερήσια διατάξη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι ίσω την επόμενη φορά θα προτιμήσετε να κάνετε το σχόλιο αυτό, ένα παρόμοιο σχόλιο κάποια άλλη χρονική στιγμή για την Τετάρτη τώρα από το, την του, της ΓΚΟΕ. Έλαβα το αίτημα για τις δηλώσεις της, ε, του Συμβουλίου για την Τουρκία το τρίτο σημείο το απόγευμα να το βάλουμε στο τρίτο σημείο μάλλον στην ημερησία διατάξη μετά τις δηλώσεις για την επαναφορά ενός ε, συστήματος Σέγγεν. Η κυρία Σπινέλη ζήτησε το λόγο για να υποστηρίξει το αίτημα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματο πολιτική μου ομάδα, θα ήθελα στην ημερήσια διάταξη να προβλέπετε μία συζήτηση σε σχέση με την Τουρκία για τα κατά πόσο πληρεί τελικά τι συνθήκε προκειμένου να καταργηθούν οι θεωρήσει την Δετάρτη ω τρίτο σημείο το απόγευμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να αναλύσουμε το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια τέτοια απελευθέρωση των θεωρήσεων, χωρί όμω να υπάρχουν οι απαραίτητε διασφαλίσει, ότι δηλαδή πληρούνται όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιο, πώς θα αναθεωρηθεί ο νόμος κατά της τρομοκρατίας και τι θα γίνει με το ζήτημα της Κύπρου. Να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας για τα δύο αυτά ζητήματα και είναι πολύ πιο σημαντική η συζήτηση αυτή μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν την Παρασκευή που είπε ότι δεν πρόκειται να τροποποιήσει την νομοθεσία τη κατά τη τρομοκρατία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή ότι στην Τουρκία κατηγορούνται και μάλιστα έχουν φυλακιστεί για λόγου τρομοκρατία καθηγητέ ή πολλοί άνθρωποι που ανήκουν στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς επίσης και δημοσιογράφοι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τι πρόκειται να κάνουμε εμείς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κινηθούμε υπό τις απειλές ή υπό τον εκβιασμό του Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν μας λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανάσχεση των μετασταυτικών ροών, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απελευθερώσει τις θεωρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάραμς ε, ζήτησε το λόγο για το αίτημα αυτό. Η ομάδα μου υποστηρίζει την πρόταση τη συναδέλφου από την ΚΟΕ γιατί πιστεύουμε ότι ιδιαίτερως μετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών ε, για τον πρόεδρο Βούτογλου, για την καταδίκη του Τζανκούντα και ως ε, ε, τρομοκράτη αλλά και την επίθεση κατά του Τσάντουντα. Μετά από όλα αυτά λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει σίγουρα σε κάθε περίπτωση να συζητήσουμε την κατάσταση γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δώσει την εντύπωση ούτε στην Τουρκία αλλά ούτε και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωση ότι δεχόμαστε πιέσεις και ότι ανεβόρον διαπραγματευόμαστε με την Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μέτσολα κατά του αιτήματο. Mr. President. The EPP group understands... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ΕΛΚ κατανοεί ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα για τι ομάδε όλε και για του πολίτε μα. Φυσικά και πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά πρέπει να γίνει υπεύθυνα και ε, εκτεταμένα. Η, Κομισιόν προτείν... η πρόταση τη Κομισιόν τη περασμένη εβδομάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί απομονωμένα από την ευρύτερη εικόνα που καλύπτει τον οδικό χάρτη Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία, την πολιτική μετανάστευση και την Ουκρανία και το Κωσυφοπέ σχέδιο. αυτόν όλων ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι κρίσιμο σε όλη αυτή τη διαδικασία αποφάσεων. Είναι θέματα επίμαχα και πολύ ευαίσθητα και γι' αυτό ε, πρέπει ακόμη περισσότερο να εξασφαλίσουμε ότι οι συζητήσεις μας θα είναι πολύ καλά προετοιμασμένες. Και πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ε, την αρμόδια επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και να εξασφαλίσουμε μια, ε, μια ε, ζωντανή συζήτηση ενώ θα σεβαστούμε τη διαδικασία που προβλέπετε. Ας πούμε, απόψε η Επιτροπή Λίμπε θα κάνει μια εκταμένη συζήτηση επί του θέματος, οπότε το ΕΛΚ είναι αντίθετο στην προσθήκη αυτού του θέματος σήμερα, τώρα. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ψηφίσουμε για το αίτημα. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματος της ΓΚΟΕ. Κατά. αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισατε παρακαλώ όλοι. Πέρασε. 181 ψήφοι Πέρα 92 κατά. Και έτσι λοιπόν, την Τετάρτη θα υπάρξει παράταση της Συνόδου μέχρι τις 12 το βράδυ. Η ε, κυρία Άρμς, για να μην τα μπλέξουμε τα ζητήματα, το θέμα είναι και η συζήτηση για τον, με τον κύριο Τίμερμαντς για το Σέγγεν. Ε, σήμερα πήραμε την είδηση ότι υπήρξαν πυροβολισμοί στα σύνορα μεταξύ Σλοβενίας και Ουγγαρία και ότι υπήρχαν και τραυματισμένοι μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, μια πρόσφυγα. Θα ήθελα στο σημείο λοιπόν αυτό να προτείνω και εσείς και στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώσετε τον κύριο Τίμριμαντς ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό στο Κοινοβούλιο το περιστατικό αυτό στην συζήτηση που θα γίνει να χτυχτεί, να σχολιαστεί και από αυτόν. Νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται για ένα σημείο να σε ό,τι αφορά ε, το Σέγγεν, αυτό που συνέβησε σήμερα στα σύνορα μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβενίας. Okay. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Για το πρόγραμμα εργασίας ε, δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο και έτσι λοιπόν αποφασίζεται η ημερήσια διάταξη έτσι. Να περάσουμε τώρα στις, ε, στην κοινή συζήτηση για την πολιτική συνοχή. Έκθεση Γιώτοβα. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Γιώτοβα.